So, ich Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ όλοι συνάδελφοι. Έχουμε μια μικρή ψηφοφορία πρώτα και μετά θα υποδεχτούμε τον Επίτροπο κύριο Μπόρτς. Λοιπόν, στο σημείο 10 ψηφίζουμε τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων και τα λοιπά, έκθεση Ζανώνη. Έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Μάλιστα. Εισηγητής, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Πρόκειται για την τροποποίηση, όπω είπατε, τη οδηγία σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Ξέρετε επίση ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, τέσσερι ή τριμερεί διάλογοι. Καλή συνεργασία είχαμε με τους κοιόδησηγητές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα λοιπόν του Κοινοβουλίου κατάφερε να καταλήξει σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μπορέσαμε να βελτιώσουμε την ισχύουσα οδηγία, αυξήσαμε τα όρια και τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η νέα οδηγία θα είναι πιο διαφανής, πιο αποτελεσματική, ε, λαμβάνει υπόψη τις νέα στοιχεία όπως η κλιματική αλλαγή και έχουμε και κυρώσεις αποτρεπτικές σε περιπτώσεις παραβάσεων και μεγαλύτερη πληροφόρηση ε, σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε μέτρα αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε όλες τις προτάσεις της ε, Ολομέλειας του Οκτωβρίου. Ε, υπήρξε ανασταλτική μειοψηφία στο Συμβούλιο που δεν μας επέτρεψε να εγκρίνουμε τα παραρτήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ούτε ξαναμπήκε το θέμα του σχιστολιθικού αερίου. και κινδυνεύουν να στείλουν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μήνυμα στην κοινή γνώμη που περιμένει απολύτως να κάνουμε κάτι. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν ε, αποφάσεις με τα λόγω γνώσεως για 200 διαφορετικά είδη έργων ε, δημοσίων και ιδιωτικών. Θα μπορέσουμε να περάσουμε πλέον αυτό το κείμενο, να το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ και ε, τους ε, υπευθύνους της Γραμματείας για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. 46 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία για την αντίρρηση σχετικά με τα νανοηλικά. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Έχετε όλο τον κατάλογο ψηφοφορία σας μπροστά σας. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά και πάλι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Υπεράριθμος ένας σοσιαλιστής και δημοκράτης. Τώρα είμαστε εντάξει, 32 υπέρ, 20 κατά, χωρίς αποχές. Το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά πάντα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρας. 34 υπέρ 22 κατά. Εγκρίνεται και αυτό. Συνολική τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. 31 υπέρ, 23 κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt 13, Angabe des Auslands bei Fleisch, das in Vorbereitung. Σημείο 13. Επισήμανση της χώρας προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται στα μεταποιημένα προϊόντα. Ηλεκτρονικά και πάλι. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 45 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Και τώρα καταφθάνει ο κύριος Επίτροπος.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 Παρακαλώ πολύ αν γίνονται διαπραγματεύσει μεταξύ φιλελευθέρων και σοσιαλιστών. Ασταματήσουμε σταματήσουμε για λίγο γιατί εδώ θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον Επίτρομο Μπόρτς για την κλωνοποίηση των ε, ζώων και φυσικά έχουμε το θέμα της ε, νομοθετικής πρότασης Έχουμε συζητήσει για το ποια είναι επί του ουσίας αρμόδια επιτροπή, ποια είναι η επιτροπή που θα πρέπει να αναλάβει το θέμα. Βλέπετε εδώ πόσοι είναι οι συνάδελφοι που είναι παρόντες εδώ. Έχουμε ένα κατάλογο ομιλητών ο οποίος είναι ήδη πολύ φορτωμένος, αλλά βεβαίως καταρχήν θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να σας εξηγήσω τους ε, λόγους πίσω από την πρόταση που υιοθέτησε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο. Όπως ξέρετε δεν υπάρχει η πρόταση που αφορά την κλωνοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν όσον αφορά την πρόταση αυτής της πρότασης. Η πρώτη όσον αφορά την απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων, όσον αφορά καταρχήν το θέμα των διάφορων ζώων, των χείρων, των αλόγων για λόγους αναπαραγωγής, αλλά και για την τοποθέτηση της, στην αγορά κλωνοποιημένων ζώων ή εμβρίων κλωνοποιημένων. Η δεύτερη πρόταση αφορά μια εμπειρία όσον αφορά το σταμάτημα της τοποθέτησης στην αγορά στην τροφική αλυσίδα. Τρόφιμα δηλαδή. Πρόκειται δηλαδή για τρεις απαγορεύσεις. Απαγορεύση κλωνοποίηση, θέτηση αυτών των ε, κλωνοποιημένων προϊόντων στην ε, αγορά και στην ε, τροφική αλυσίδα. Αφού υιοθετηθούν και εγκριθούν αυτές οι προτάσεις, ακολουθήσουν οι εκθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των οδηγιών. Και εδώ βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας ε, και την τεχνική πρόοδο, την επιστημονική πρόοδο, αλλά και την ε, εξέλιξη στα κράτη-μέλη. Γιατί καταρχήν αυτή η απαγόρευση της κλωνοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν θέματα εφημερίας των ζώων. Το θέμα της ε, κλωνοποίησης αυτής και θεαυτής, αλλά και της φέρουσας μητέρας, και βεβαίως όσον αφορά το θέμα της ε, ε, της μητέρας και του κινδύνου για την ε, υγεία της, τους θανάτους που προκαλεί. Υπάρχουν βεβαίως σήμερα σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την κλωνοποίηση για την παραγωγή ε, τροφίμων και πολλά κράτη-μέλη βεβαίως έχουν υιοθετήσει με τέτοια απαγόρευση εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί εγγράφως τον Οκτώβριο του 2013 στον Πρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Μπαρόζο, και στις 29 Μαρτίου του 2011 ξεκίνησε στο Συμβούλιο η πρόταση όσον αφορά την σήμανση ε, νοπού κρέατος που προέρχεται από κλωνοποίηση. Επίσης, η Επιτροπή σας έχει εκφράσει την άποψή όσον αφορά τη σήμανση τροφίμων <clears throat> που περιέχουν κλωνοποιημένα Μετά την αποτυχία της συνδιαλλαγής το 2011, η Επιτροπή είχε υποσχεθεί ότι θα ε, προετοιμάσει μια ξεχωριστή νομοθεσία για θέματα κλωνοποίησης και βεβαίως σε σχέση με τις αρμοδιότητές μας και σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας μία περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης, όταν εξετάσαμε δηλαδή διάφορες εναλλακτικές, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τη σήμανση των τροφίμων. Και αυτό βεβαίως ήταν κάτι που σαφώς και μας δημιουργήσε προβλήματα όπως προβλήματα ίχνηλασιμότητας. Εγώ όταν παρουσίασα την πρόταση αυτή, βεβαίως έδωσα και μία τρίτη εναλλακτική όσον αφορά τη σήμανση. Και μία από αυτές ήταν και το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε να εξετάσει αυτές τις τρεις τις εναλλακτικές. Όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ε, ζώα, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται ειδικέ και επιπλέον πληροφορίες για κάθε ε, τέτοιο προϊόν, κάτι που φυσικά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα για κάθε επιπλέον γενιά κλωνοποιημένων ζώων. Κάτι που φυσικά αυτό συσσωρεύεται και γίνεται πιο περίπλοκο για την κάθε επιπλέον γενιά. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι όλη η παραγωγή, κτηνοτρόφοι, ειδικά θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτήν την αλυσίδα που απορρέει από την κλωνοποίηση και αυτό βεβαίως ε, η επιπλέον ανάγκη συσσόρευσης πληροφοριών και σήμανση αυξάνει σημαντικά και το κόστος τελικά του τελικού προϊόντος. Το θέμα είναι βεβαίως γιατί ακριβώς ε, επιπλέον κόστος ε, πρόκειται. Γιατί αυτό επηρεάζει και το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης. Και βεβαίως εξετάζοντας αυτές τις τρεις εναλλακτικές θα έλεγα ότι καταρχήν, όπως ανέφερε και η ΕΦΣΑ, η Υπηρεσία Ασφάλειας των έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ε, ευημερία των ζώων, της, της μητέρας, παραδείγματο χάρη, και όσον αφορά την πρώτη εναλλακτική, δηλαδή το σταμάτημα αυτής της ε, κλωνοποίησης, της τεχνικής για την παραγωγή ε, μου βασίζεται στο άρθρο 43 με αναφορά στο άρθρο 30 της συνθήκης όσον αφορά την ευημερία των ε, ζώων. Και όσον αφορά την δεύτερη πρόταση, δηλαδή ε, τρόφιμα αποκλωνοποιημένα ζώα, πρόκειται για τρόφιμα που προέρχονται από ζώα και εκεί δεν υπάρχει θέμα ε, τέτοιας ευημερίας ζώων και σε καμία περίπτωση από τη στιγμή που τα ζώα αυτά έχουν ε, παραχθεί με συμβατικές μεθόδους, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ευημερίας των ζώων. Σκοπός μας, κύριε Πρόεδρε, είναι να σταματήσουμε την εξάπλωση μιας μεθόδου παραγωγής, μιας ε, τεχνικής η οποία δεν ακολουθεί κανόνες δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να λάβουμε μια τέτοια αναλλακτική λύση υπόψη μας από τη στιγμή που η συνθήκη δεν μας επιτρέπει ούτε βάσει του άρθρου 43 ούτε του 14 που αναφέρεται στην εσωτερική αγορά, το 160 που αφορά και το 169 που αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών δεν αναφέρεται σε αυτές τις νομικές βάσεις. Άρα η 352, το 352 άρθρο που αφορά την ρήτρα της ε, ευελιξίας μπορεί εδώ να θεωρηθεί σαν βάση, δεν δίνει όμως σε καμία περίπτωση αυτή τη δυνατότητα, διότι μπορεί κανείς να τη θεωρήσει απλώς μια εξαιρετική διαδικασία, νομοθετική διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα εδώ, αναφερόμενος στην σήμανση, που δεν αναφέρεται σε αυτή την πρόταση εξάλλου, να πω ότι το σύνολο των επιτρόπων δεν αποφάσισε η σήμανση τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα γίνει είναι κάτι το δυνατόν, αλλά πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο θέμα όσον αφορά τουλάχιστον τη σήμανση νοπού κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα και θεωρεί ότι εδώ χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν ληφθεί η απόφαση αν ναι ή όχι μπορεί να θεωρηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική σήμανση σαν την ορθή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα αφού έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δε, αργότερα μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Δεν λέω δηλαδή ότι αυτή είναι η ορθή απόφαση, λέω όμως ότι ουσιαστικά η Επιτροπή αποφάσισε ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν είναι ικανή να πάρει απόφαση για το θέμα αυτό της σήμερα της ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμπέραντα βεβαίως σεβόμενη εδώ το νομικό πλαίσιο πιστεύω ότι ναι προτείνει εδώ η Επιτροπή ένα νομοθετικό πλαίσιο. Βεβαίως η άλλη νομοθετική αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί και ελπίζω ότι οι σημερινές μου επεξηγήσεις μπορεί να μην σας ικανοποίησαν πλήρως, αλλά τουλάχιστον ε, ανταποκρίνονται στη δέσμευση της Επιτροπής να κάνει μία πρόταση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δεν ξέρω αν μας ικανοποιήσετε. Τολμώ να το αφισβητήσω αυτό. Μετά την παρουσίασή σας ε, έχουν στήσει πολύ το λόγο, θα γίνει ευρία συζήτηση. Και σε ό,τι αφορά ε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου και τι θύρες ανοίγονται με αυτή την πρόταση. Θα τα ακούσετε τώρα από τους συναδέλφους σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, αρχίζουμε από τους συντονιστές όσοι ήθιστε, ο κύριος Πέτερ Λίζε πρώτος, η κυρία Μακάβαν και μετά οι υπόλοιποι ομιλητές. Παρακαλώ, Πέτερ Λίζε. Σύντομα παρακαλώ όσο γίνεται για να προκάνουμε και να πάρουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι και να κάνουν τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε αγαπητέ Τόνιο Μπόρτς. Είναι πραγματικά θαραλέο που έρχεστε να παρουσιάσετε αυτό το θέμα ενώπιον της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ για το θάρρος σας και το κουράγιο και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που φέρατε εγκαίρως την πρότασή σας. Την είχατε εξαγγείλει για πέρυσι βέβαια και ξέρω ότι η εσωτερικά της υπηρεσία σας ήταν αμφιλεγόμενη, εν πάση περιπτώσει ήρθε. Και γνωρίζω ότι αγωνιστήκατε και εσείς προσωπικά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου περισσότερο. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά και να σας συγχαρώ, αλλά παρακαλώ κατανοήσετε ότι είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι στην Επιτροπή μας ε, που ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολείπεται κατά πολύ των όσων περιμέναμε. Λιγότερα από αυτά που το Συμβούλιο και το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν φέρει στο Κοινοβούλιο ε, στις διαπραγματεύσεις και το επιχείρημα ότι χρειάζεται περαιτέρω διευρεύνηση δεν πιάνει. Δυόμιση χρόνια το κουράζεται πριν από δυόμιση χρόνια είχαμε περισσότερα ε, να προσφέρουμε και τώρα μας λέτε χρειάζονται νέες έρευνες. Το θέμα της επισήμανσης των επομένων γενναιών ζώων, ε, αν μπορεί να γίνει αυτή, ε, το μελέτησα πάρα πολύ εντατικά, το έχω κοιτάξει γιατί ξέρετε ότι είμαι γιατρός και έχω εργαστεί στην ανθρώπινη γενετική, έχω κάνει το διδακτορικό μου και την υφηγησία και με εταιρείε που κάνουν τεστ DNA. Έχω συζητήσει και έχω ρωτήσει, είναι δυνατόν όταν έχει ένα κλωνοποιημένο ζώο ε, να έχει απογόνους και προϊόντα, χρειάζεσαι μήνες ε, για να το μελετήσεις και να έχεις το αποτέλεσμα. Ε, αυτά που μας λέτε δεν ευσταθούν. Οι δικοί μου έχουν πει τα αντίθετα και θα παρακαλούσα ε, να το κοιτάξετε. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Η συμφωνία TTIP ελευθέρων συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείες έπαιξε ρόλο στη συζήτηση από ό,τι άκουσα και αν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτή τη συμφωνία ε, μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών για να μην ε, καταρρεύσει η συμφωνία. Ας καταρρεύσει η συμφωνία. Υπάρχει ένα θέμα με τη στρατηγική διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το καλοκαίρι που είχαμε πάει με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες η αρμόδια για το εμπόριο του Προέδρου Ομπάμα και της FDA, της Υπηρεσίας για τα Τρόφιμα και τα ε, φάρμακα μας είπαν «Ε, μα να διαπαιδαγωγείτε καλύτερα το λαό σας. Έχουν παρέλθει αυτοί οι καιροί. Εμείς δεν είμαστε αναμορφωτήριο να διαπαιδαγωγούμε τους λαούς μας. Εκπροσωπούμε τους πολίτες που μας έχουν εκλέξει. Να τα πούμε αυτά στους Αμερικανούς. Και ένα τελευταίο. Οι κρατικές αρχές με ρώτησαν διαφόρων κρατών μελών. Γιατί όλο αυτό είναι οδηγία. Αφού είναι δύσκολη η εφαρμογή, καλό δεν θα ήταν να υπάρχει ε, μια σαφήνεια για το πώς θα εφαρμοστεί. Και είναι ένα αίτημα το οποίο εγώ διαβιβάζω και μόνο μήπως μπορεί να γίνει οδηγία κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ για τα δύο λεπτά που τηρήσατε κύριε Λίζε, δεξής τρισήμιση, Η κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ. Ήμουν τμήμα της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας στον τριμερή διάλογο. Και ο λόγος που το Κοινοβούλιο είπε όχι τότε είναι γιατί θεωρούσαμε ότι είχαμε μία άτιμη πρόταση, για να το πω έτσι. Ε, επαναλάβατε τώρα αυτά που ξέραμε, ότι η Επιτροπή Διαντολογίας είπε ότι είναι ανήθικοι, ότι υποφέρουν τα ζώα. Και όμως η Κομισιόν είναι, ήταν τότε έτοιμη και ακόμα και σήμερα ετοιμάζεται να επιτρέψει την εισαγωγή α, κλωνοποιημένων υλικών και ούτε καν τα επισημαίνει αυτά. Ξεκινήσαμε με την εισαγωγή α, σπέρματος από τη Σκοτία. Ε, ε, τότε λέγαμε είναι νόμιμο ή όχι, είχε σταματήσει, αυτά είχαν γίνει. Τώρα λέει τι λέμε. τα κλωνοποιημένα ζώα, ας πούμε, τα, τα επιτρέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπουμε ε, να τα κλωνοποιούν και εμείς εισάγουμε, ας πούμε, το, το σπέρμα, τα εισάγουμε μετά και έχουμε, πλήπτουμε τα σχήρας. Ε, έχουμε εμείς ψηλά πρότυπα. Τα αφήνουμε σε αυτούς. Δεν νομίζω είναι σωστό αυτό. Και όπως είπε και ο Πίτερ Γκλίσε, η Κομισιόν είχε πει πριν από δύο-τρία χρόνια ότι θα μπορούσε να υπάρξει ίχνη είχε κάνει κάποιες ταπεινές προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και τώρα μας λέτε καμία επισήμανση. Είναι απαράδεκτο. Και για να είμαι και λίγο κοινική θα σας έλεγα ότι το Σώμα των Επιτρόπων το σκέφτηκε κάποτε χωρίς καμία επισήμανση. Στην πραγματικότητα θα το περάσετε μέσω της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων. Δεν θα μας, θα μας παρακάμψετε εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας που έχουμε πολύ στεναρές απόψεις γι' αυτό. Ε, Όμω υπάρχει μια ε, διαπαραταξιακή συνένεση για το πώ πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα και διαφωνούμε κάθετα με την πρόταση τη Κομισιόν. Λυπάμαι. Η κυρία Κορίν Λεπάζ, ε, εξ ονόματος Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, ε, Επίτροπε, που ήρθατε. Εγώ θα είμαι ακόμα πιο έντονη. Όπως η κυρία Μακάβαν και εγώ είμαι τμήμα τη της διαπραγματευτικής στον Τρίγλογο και Ήμασταν πολύ υποχωρητικοί σε σχέση με αυτά που θέλαμε αρχικά, που ήθελε, με αυτά που ήθελε το Κοινοβούλιο και ο ευρωπαϊκό πληθυσμό. Ε, Κανένα δεν θέλει να καταναλώνει ζώα από ε, από κλωνοποιημένα ζώα. Ε, μας λέτε ότι κοστίζει ακριβά. Το θέμα δεν είναι τεχνικό. Ε, Σα το είπε και πολύ καθαρά ο Πίτερ Λίσε. Το θέμα είναι πολιτικό τελικά, Επίτροπε. Και με διπλό τρόπο. Από τη μία στην έκθεση, ε, στη σχέση μεταξύ Ευρώπης, είπα, στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλογών. Τι μας προτείνεται, να χαμηλώσουμε τον πύχη πριν ξεκινήσουμε καν τις διαπραγματεύσεις και να δεχτούμε ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, να μειώσει τα πρότυπα ασφάλειάς του και τα πρότυπα ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτό. Επίσης υπάρχει και πρόβλημα δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο. Θα ξέρετε φαντάζομαι την αμηχανία που προκλήθηκε μετά από τη χθεσινή συζήτηση στο Συμβούλιο για τους ε, γάματα φόμικρων. Οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν, παρά την αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά την αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών μελών, να επιτρέπουμε τους γενικά, γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς ε, και να συζητάτε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και για τους κλωνοποιημένους και τα κλωνοποιημένα τρόφιμα το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Τι θέλουμε, και το θέση. είναι δικαίωμα του Ευρωπαίου καταναλωτή. Το έχει κατακτήσει. Και τι μας προτείνετε εσείς, να αγνοήσουμε αυτό το δικαίωμα, δεν το δεχόμαστε, δημοκρατικός πώς είναι απαράδεκτο, εδώ εκπροσωπούμε τους ευρωπαϊκούς λαούς, το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων, δεν θέλουμε να γλύψουμε την α ή β ε, βιομηχανία αγροτροφίμων και επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε επίτροπε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, Παρτιστάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Απογοήτευση, τι να πω. Εντάξει, ακούτε τώρα. Έλεγα λοιπόν, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταλαβαίνετε, Επίτροπε, ποια είναι η απογοήτευσή μας, ακούσατε τις προλαλήσαντες από τις τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω κι εγώ με κάποιους συναδέλφους εδώ πολύ καιρό διαπραγματευόμαστε για τα νέα τρόφιμα, Novel Food, πήγε μετά στην κλωνοποίηση, νύχτες ολόκληρες στο Συμβούλιο και τώρα αυτό που μας προσφέρεται υπολείπεται κατά πολύ. Η χνηλασινομότητα, τα είπαν και οι συνάδελφοι, ήδη από το 2010 είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι δυνατόν και από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοί σας, οι επίτροποι, είναι πολύ πιο ισχυρή από τις δικές της υπηρεσίας που γνωρίζουν περισσότερα και υποθέτω ότι και εσείς είστε στο δικό μας πλευρό. Ο κύριος Λίζε ε, ε, ε, με βρίσκει σύμφωνο. Για την επισήμανση και την ετικετοθεσία είναι εκ των όνων κάνευ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει κάποια ρύθμιση. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ ε, των θεσμικών οργάνων στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό νέα τρόφιμα, novel food, και τώρα υπαναχωρήσατε. Ε, χρησιμοποιήθηκαν πολλά επιχειρήματα. Ε, όχι μόνο η επιμερία των ζώων και ε, άλλης φύσεως. Συμφωνώ με τους υπολείπους συναδέλφους. Τι γίνεται στο κολέγιο των επιτρόπων. Υπάρχουν και ε, θέματα διεθνούς εμπορίου που έπαιξαν ρόλο και ένας φόβος ότι μην τυχόν και δεν μπορέσουμε να κλείσουμε τη συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μήπως τώρα Έχουμε περάσει κάτω από τον πύχη γιατί παίζουν άλλα πιο σημαντικά ζητήματα. Όλη η οδηγία για την κλωνοποίηση περιορίζεται σε συγκεκριμένα είδη ζώων, κάποια άλλα εξαιρούνται και είναι μόνο για σκοπούς ε, γεωργικούς. Ας πούμε, όχι ζώα που γίνονται πειράματα επιστημονικά. Και ε, τελευταίο είναι και οδηγία. Και μάλιστα μία από τις οδηγίες που δεν είναι και σε συναπόφαση. Τι ωραία. Πραγματικά νομίζω μας περιπέζετε, ε, θέλετε να μας παραγωνίσετε και είμαστε πολύ απαγοητευμένοι με αυτά που έχει φέρει η Επιτροπή ως πρόταση και προτιμούμε φυσικά κανονισμό από δίγεια. Ευχαριστώ κυρία Καρτίκα Λιωτάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη είπαν οι προλαλήσαντες για το εμπόριο, αλλά με λίγο που ήρθατε εσείς να μας κάνετε αυτή την πρόταση και να την περασπιστείτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πιστεύω ότι τα έχει μαγειρέψει ο κύριος Ντεχόχτ αυτά, όχι εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς τολμάτε να μας πείτε ε, ότι είναι η δική σας πρόταση. Υποθέτω ότι έχετε ακούσει ε, πολλά για δεοντολογία, για ασφάλεια τροφίμων, για την ευημερία των ζώων. Γνωρίζετε ότι 70% του πληθυσμού δεν συμφωνεί με την κλωροποίηση ε, ζώων για σκοπούς ε, διατροφικούς και μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά τα παράπονα στον κύριο Ντεχούχτ παρακαλώ. Γνωρίζετε ότι το κρέας και άλλα προϊόντα προέρχονται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, όχι από το ίδιο το ζώο που έχει κλωνοποιηθεί. Και διερωτώ με, γιατί ε, δεν ε, συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή σας. Κατά την άποψή μου θα πρέπει ε, να απαγορεύεται, ας πούμε όπως απαγορεύεται να έχουμε αυγά που τα έχει γεννήσει ένας κόκορας, διότι τα κοκόρια δεν γεννούν αυγά και τα κλωνοποιημένα επίσης δεν γεννούν. γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαγορεύει την ε, παραγωγή τροφίμων από απογόνους κλωνοποιημένων. Για μη τι άλλο να υπάρχει μια ετικέτα και να γνωρίζει ο καταναλωτής τι τρώει. Εγώ είμαι υπέρ της απαγόρευσης. Ε, θα μπορούσα να συμβιβαστώ και με ε, την ετι, και το θεσία και τη σήμανση και μπορείτε να μας εξηγήσετε παρακαλώ γιατί χρειάζεται τέσσερα χρόνια για να φέρετε αυτή την πρόταση. Ένα νομικό τέχνασμα φέρετε στο κοινοβούλιο για να βγάλετε off-site στο κοινοβούλιο. Σας χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια γι' αυτό. Και λέτε ότι είναι το άρθρο 352 της Συνθήκης Λισαβόνα νομική βάση αντί του συνήθους 114 γιατί κυριάρχησαν οι σκέψεις της αγοράς και του εμπορίου. Για να μην έχει καμία δυνατότητα το Κοινοβούλιο να κάνει τίποτα. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχολείται και με την ουσία του θέματος όσο ασχολείται με το να επινοήσει διάφορα νομικά τεχνάσματα για να μας παρακάμπτει. Παρακαλώ να αποσύρετε την πρόταση και να φέρετε νέα βάση του άρθρου 114 της συνθήκης και θα είμαστε εντάξει εάν σε αυτή την πρόταση τελικά είναι στο προσκήνιο το συμφέρον και η επιθυμία του καταναλωτή, ο οποίος να ξέρει και τι θα τρώει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο θα έχει ο Επίτροπος, ο κύριος Μπότς, για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων, των συντονιστών. Και μετά έχει και άλλο γύρο. Okay. ECR group, chairman. Yeah. Ε, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές έχουν και αυτοί συντονιστεί. Εγώ θα χαλάσω την ωραία συνένεση εδώ πέρα που υπάρχει, υποστήριζοντας την Κομισιόν. Καταρχάς, θέλω να πω στη Λίντα Μακάβαν ότι δεν ήταν σπέρμα από κλωνοποιημένο ζώο της σκοτίας που στα εστάλθη στην Αγγλία. Ένας ακτινοτρόφος ε, εισήγε από την Αμερική. Ε, έσφαξε το τάβρο στη Σκοτία και το κρέας έφτασε στις Βρυξέλλες. Και παρόλα αυτά στις Βρυξέλλες δεν υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί στους δρόμους. Καταναλώνουμε ε, ε κρέας από τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων από την Αμερική εδώ και χρόνια. Ακόμα και σε αυτή, τη, αυτή χώρα εδώ, για χρόνια. Η Κομισιόν μας είπε ότι η ΕΦΣΑ λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των τροφίμων. Αν μιλάμε για εισαγωγή απαγόρευσης, ενώ στην Αμερική δεν έχουν καμία τέτοια απαγόρευση στην ε, κλωνοποίηση, δεν έχουν τα καθόλου, και τότε θα αρχίσει ένα εμπορικό πόλεμο εδώ πέρα, που θα ματώσουν πολλές μύτες. Καμία σχέση με τον πόλεμο της μπανάνας πριν από 10 χρόνια. Θα είναι μια τελείως ε, άλλη ιστορία, πολύ πιο σκληρός. Εκείνος ο πόλεμος θα μοιάζει με πόλεμο μωρών. Όλοι λέτε εδώ πέρα ότι εκπροσωπείτε τους πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν κλωνοποίηση. Εγώ μίλησα με χιλιάδες πολίτες ω Ευρωβουλευτή. Κάθε χρόνο το κάνω μάλιστα. Και ούτε ένα από αυτού δεν μου είπε ποτέ ότι το να απασχολεί το θέμα τη κλωνοποίηση. σω οι Σκοτσέζοι δεν έχουν πρόβλημα τέλο πάντων με την κλωνοποίηση. Αλλά ούτε ένα ε, δεν το είπε. Και αν οι έσα που είναι εμπειρογνώμονε λένε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλεια, τότε εντάξει, να απαγορεύσουμε την κλωνοποίηση, αλλά να επιβάλλουμε οπωσδήποτε την επισήμαση είναι απαράδεκτο. Και εγώ υποστηρίζω την Κομισιόν και το Σώμα των Επιτρόπων που υπερασπίζεται την, ε, τις αρχές της και λέει δεν θέλουμε ρε παιδί μου κλωνοποίηση, ε, συγγνώμη, επισήμαση. Ο Επίτροπος τώρα, παρακαλώ. Ορίστε. Ακούμε δύο ε, άτομα που δεν συμφωνούν μαζί μας πολιτικά και όμως λένε ότι είμαστε θαραλέοι. Δεν θέλουμε τώρα εμείς να φυσικάσουμε βέβαια, έτσι. Γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πριν να αποφασίσουμε οριστικά. Αλλά ας ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για αυτό το θέμα. Αν υπάρχει διάταξη επισήμασης ή αν υπάρξει, δεν θα υπάρξει για λόγους ασφάλειας. Αν είναι κάτι μη ασφαλές, το απαγορεύουμε. Δεν το ρυθμίζουμε με επισήμανση. Αν είναι μη ασφαλές, επικίνδυνο δηλαδή, το απαγορεύουμε. Αν μία υπηρεσία, ένας οργανισμός, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίνει επιστημονική συμβουλή για θέματα ασφάλειας, τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο επίτροπο. Πρέπει να χρησιμοποιεί μερικέ φορέ την εύσα και μερικέ φορέ να την αγνοεί. Όταν μιλάει για την απαγόρευση των, της νοικοτήνης ας πούμε, και των προϊόντων νικο, γιατί δεν είναι καλό για, την, για τον πληθυσμό, να συμφωνήσω τότε. Και όταν, είναι, ε, όταν μια απόφαση της ΕΦΣΑ ή μια συμβολή της ΕΦΣΑ είναι πολιτικά ε, μη δημοφιλής, τότε την αρνούμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να την ε, χρησιμοποιούμε την ΕΦΣΑ à la carte, όποτε μας βολεύει. Παραδείγματο χάρη. Ε, Εμεί δεν θέλουμε, α πούμε, οι τρίτε χώρε να παίρνουν πολιτικέ αποφάσει και να μπλοκάρουν κάποιε από τι εξαγωγέ μα. Και ενώ καταγγέλουμε αυτή την πολιτική στάση των τρίτων χωρών, εμείς οι ίδιοι να την χρησιμοποιούμε και να την υιοθετούμε. Όταν το θέμα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων. Θα ήταν αντίφαση αυτό. Ε, να πούμε, ας πούμε, εντάξει, θα το επισημάνουμε γιατί είναι ε, μη ασφαλές. Υπάρχουν επιχειρήματα. Εγώ τα υπέβαλα στο Σώμα των Επιτρόπων υπέρ ή κατά της επισήμασης. Φυσικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επισήμαση ε, φρέσκου βοήου πρώτης γενιάς και την επισήμανση των επομένων γενναίων. Φυσικά υπάρχει και διαφορά στο κόστος ανάμεσα στην επισήμανση ενό είδου κρέατος ή όλων των ειδών κρέατος. Φυσικά υπάρχει διαφορά κόστους. Αυτό που υπέβαλα στους επιτρόπους ήταν οι διάφορες επιλογές που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επισήμανσης, για το θέμα της επισήμανσης. Επαναλαμβάνω, οι επίτροποι δεν είπαν κλείνουμε την πόρτα στο θέμα της επισήμανσης, είπαν είναι περίπλοκο, πρέπει να το μελετήσουμε και μπορεί στο μέλλον να δεχτούμε κάποιες προτάσεις που να αφορούν την επισήμανση. Αλλά σε αυτή τη φάση αυτό δεν είναι δυνατό. Και ένα άλλο επιχείρημα τώρα. Μπορούμε να έχουμε επισήμανση επί κάποιου πράγματος όπου η ανιχνεσφημότητα βασίζεται μόνο σε έγγραφα. Θα ήταν καλύτερο να είχαμε και επιστημονικές δοκιμές, αλλά έχουμε ειδικά περιπτώσεις όπως στα παράγωγα γαματαθόμικρων όπου η επισήμανση ε, βασίζεται σε ανιχνευσιμότητα η οποία βασίζεται στα έγγραφα μόνο. Φυσικά, αν θέλαμε επισήμαση και στο γάλα θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερε δυσκολίε γιατί έχουμε μείγματα α, γάλακτος αποκλεινοποιημένα και ζώα. Επίσης, μου θέσατε το ερώτημα για το TTIP. Εδώ επίσημα δηλώνω ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση και από τις δύο πλευρές να φτάσουμε συμφωνία. Όντω, το λέω. Είναι σαφέ ότι η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στην Κομισιόν είναι, τη δείχνουμε γιατί. Για να βρει λύσεις στα προβλήματα. Όχι προβλήματα στις λύσεις, αλλά το κάνουμε όχι θυσιάζοντας τα πάντα. Και το τι το δεν ήταν ε, το βασικό μας μέλημα για να αποφασίσουμε αν θα συμπεριλάβουμε τις διατάξεις ε, επισήμασης ή όχι. Γιατί σε ό,τι αφορά τον οπό βόλιο, όταν υπάρχει εξαγωγή από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, τα κανάλια είναι διαχωρισμένα ε, στις εξαγωγές. Δηλαδή, μπορούμε να εξάγουμε γαλακτοκομικά χωρίς πρόβλημα με την τύπη. Τι τύπα. Επίσης με ότι έχουμε νομοθεσία γάματα αφόμικρον, γιατί επιτρέπουμε τα γάματα αφόμικρον. Αν τα απαγορεύαμε, δεν θα χρειαζόμαστε νομοθεσία. Έτσι. Γιατί έχουμε επισήμαση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Γιατί του επιτρέπουμε. Αν ήταν απαγορευμένοι, δεν είχε νόημα να του επισημαίνουμε. Και μιλάμε για νομοθεσία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που έλεγαν ότι μπορούμε να επιτρέψουμε εισαγωγή βοήου συγγνώμη, ε, εισαγωγή γάματα φόμικρο και να επιτρέψουμε και την καλλιέργειά τους. Κυρία λεπάσ, γιατί προτείνουμε μία πρόταση την οποία επέτρεψε το Κοινοβούλιο για να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν από μόνα τους αν θα επιτρέψουν την καλλιέργεια των γάματα αφόμικρων στο έδαφος τους και παρότι υπάρχουν 25 κράτη-μέλη υπέρ και ένα κατά, μπλοκάρεται. Και εγώ να σας πω, ε, μου κάνει εντύπωση που είναι έτσι τα πράγματα. Σας απαντάω για το θέμα του 1507, για τους γράμματα αφόμικρων. Καλώς. Και τώρα έχουμε τις εξής συναδέλφους. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο και μετά θα κλείσει όμως ο κατάλογος. Α, να προσθέσω κάτι, λέει ο Επίτροπο, συγγνώμη που ξέχασα. Ναι, όσον αφορά τη νομική βάση, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με τη νομική βάση, ούτε κάτι που κρύπτεται όπιστε. Και αυτό σε μία συγκεκριμένη πτυχή που είναι, αν θέλετε, το θέμα της αγοράς. Εγώ προσπάθησα την ε, νομική βάση του άρθρου 114. Θα μου άρεσε πολύ περισσότερο αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το 114 για τους λόγους που αναφέρατε. Συμμετοχή του Κοινοβουλίου δεν θα ήταν η ίδια. Όμως, όμως, με το 114 και μετά από τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί είναι τεχνικό το θέμα, είναι τεχνικό το θέμα, επαναλαμβάνω, με το 114 και σε σχέση με την εσωτερική αγορά, έχει σε σκοπό την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας, ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αγορά κλωνοποιημένων ζώων ή ε, τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από γόνους κλωνοποιημένων ζώων και δεν υπάρχει θέμα στρέβλωσης αυτής της αγοράς. Άρα η προϋπόθεση, αν θέλετε, για την νομική βάση του άρθρου 114 δεν πληρούνται εδώ. Αυτή είναι η γνωμοδότηση που μου έδωσε η νομική υπηρεσία. Από πολιτικής απόψεως θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, πρέπει να τηρήσω αυτή την γνωμοδότηση. ich Έχασα κάποιον. Όχι. Ολοκληρώνεται λοιπόν και ο κατάλογος των ομιλητών. Σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να προτείνω να περιοριστούμε σε ένα λεπτό χρόνο ομιλίας. Αλλιώς δεν θα έχουμε απάντηση. Εντάξει. Πολύ λογική. Τι μπορεί κανείς να πει σε ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, δεν θα αναφερθώ στην νομική βάση γιατί δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσατε να είσαστε πολύ πιο τολμηροί εσείς και η υπηρεσία σας, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να αναφερθώ εγώ και θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. Δεν αναφερόμαστε εδώ στην ασφάλεια των ε, τροφίμων. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχει σωστές ε, αξιολογήσεις. Εδώ όμως μιλάμε για το πώς η κοινωνία μπορεί να αποδεχθεί αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων. Όσον αφορά τα novel foods και όσον αφορά τα καλλιτικά, πριν από πολλά χρόνια, 15 και 10, ξέρετε ότι συζητήθηκαν τα θέματα αυτά και είχαμε ακριβώς την ίδια, ε, το ίδιο θέμα όσον αφορά την αποδοχή από τους πολίτες, από την κοινωνία. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιο εδώ ότι ναι, τα κλωνοποιημένα ζώα πραγματικά μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Αλλά εδώ στρέφουμε στον κύριο Στίβεν και θα έλεγα ότι κάτι το οποίο προκαλεί τον καρκίνο δεν μπορεί να εισαχθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το ίδιο θα έλεγα και για τα κλωνοποιημένα ζώα και για τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Δεν θέλουμε την εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη και πραγματικά αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούμε. Ματσάι Κούκοβιτς. Κυρία Ματσάι Κούκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπόρζ, σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ένα λεπτάκι έχω. Οπότε θα πω μόνο το εξής. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολύ ψηλές τεχνολογίες, και η γενετική και η ιατρική μας ξεπερνάει από δεξιά και από αριστερά. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει πια και τι δεν υπάρχει. Σήμερα μάθαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανάπτυξης ότι η διαχείριση των δεδομένων είναι σήμερα το πιο σημαντικό πρόβλημα. Είναι ε, ε, τεράστιος ο αριθμός των ε, ερευνητών που ασχολούνται μόνο με αυτό. Λοιπόν, για τη συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε, θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την κλωνοποίηση, ποια είναι τα ε, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και την υγεία στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ κυρία Μορκουνάιτε για ένα λεπτό. E, e, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή. Συζητάμε τα κλωνοποιημένα ζώα σήμερα, αλλά θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση λιγάκι διαφορετική που αφορά κάποια πράγματα που έχουν σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική γρήπη. Μερικά κρούσματα εμφανίστηκαν στη χώρα μου που προέρχονταν όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από τη Λευκολοσία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία άρχισαν να περιορίζουν ε, τις εισαγωγές χείριου από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το δυσανάλογο μέτρο της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μπορείτε να το σχολιάσετε. Έχετε κάποια θέση. Ίσως υπάρχουν κάποιες εξελίξεις για αυτό το θέμα. Και τι βοήθεια θα μπορούσε να περιμένει η Λιθουανία για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί ένα από τα μέτρα είναι η σφαγή ας πούμε των ζώων, αλλά αυτά είναι πολύ δαπανηρά μέτρα, πολύ ε, ριζικά μέτρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Κοιτάμε ε, αυτή τη στιγμή τα κλωνοποιημένα ζώα, αυτά καθε και όχι τους απογόνους τους. Αγνοείτε τον Ευρωπαίο πολίτη, έτσι πως μιλάτε. Αν ο Ευρωπαίος πολίτης έχει πρόβλημα με την ευμερία των ζώων, με τα δικαιώματα των ζώων και δεν θέλει να τα φάει, ε, μάλλον ε, έχει πρόβλημα και με την παραγωγή τους. Λέτε ότι θέλουμε να, θέλετε να επισημαίνετε τα κλωνοποιημένα, αλλά όχι τους απογόνους τους. Αν λέτε κάτι τέτοιο, μπορώ να πω ότι είναι γελίο. Γιατί δεν είναι σοβαρό, σοβαρό αυτό το επιχείρημα. Και μετά από τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, ε, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στη Herald Tribune που έλεγε ότι υπάρχουν διάφορα κράτη-μέλη τα οποία έχουν κλαδικά συμφέροντα Είπαν οι Αμερικάνοι. Μπορούμε να κοιτάξουμε αυτά τα κράτη-μέλη και τα, τα επιχειρήματά τους. Πρέπει να δούμε τα συμφέροντα που υπησέρχονται εδώ για να ξέρουμε τι συζητάμε. Και να μην τα συζητάμε έτσι γενικά και αόριστα και αφηρημένα. κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η κυρία Ροτ δεν αμφισβητούμε εδώ τις αξιολογήσεις της ΕΦΣΑ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά 81% οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι δεν έχουν λυθεί υπόψη ακόμα ούτε καν οι επιπτώσεις, οι μακροχρόνιες ε, επί του περιβάλλοντος, ότι μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και ότι σίγουρα η χρησιμοποίηση κρέατος, ε, τροφίμων από ζώα δεν μπορούν σήμερα να εκτιμηθούν σωστά. Και εδώ αναφέρομαι και στα προϊόντα και κατευθείαν από τα κλωνοποιημένα ζώα αλλά και από τους απογόνους τους. Υπάρχει μία απόρριψη. Το θέμα λοιπόν για την μη σήμανση, μη ετικετοθεσία, είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν αν τα κλωνοποιημένα προϊόντα εμπεριέχονται σε, στα προϊόντα τα οποία έχουν ε, προσπόληση. Και αυτό είναι το θέμα πολλές φορές και σε καμιά περίπτωση, περιπτώσει, δεν είναι έτοιμη η κοινωνία να δεχτεί μια τέτοια σήμανση. Σας ευχαριστώ. Εγώ εδώ θέλω να εκφράσω την οργή μου, τον θυμό μου. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε κύριε Επίτροπε να στηρίξετε μια τέτοια θέση. Οι καταναλωτές είναι αντίθετοι και όταν μας μιλάτε για εμπορικό πόλεμο δεν καταλαβαίνω. Η Ευρώπη είναι τόσο αδύναμη, θα τις επιβάλλουν ό,τι θέλουν. Αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεριφερθεί επιτέλους λίγο διαφορετικά, ιδιαίτερα όταν συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε σε μία προεκλογική περίοδο. Πώς θα εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη όταν διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται τα πάντα, είναι διατεθειμένη να δεχτεί τα πάντα. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν θέλει κλωνοποιημένα ζώα. Ευχαριστώ, η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μερικοί συνάδελφοι βλέπουν θάρρος από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ βλέπω λαζονία από πλευρά της Επιτροπής και από ένα τμήμα του Συμβουλίου απέναντι στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θυμίζω έχει εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες θα δεχτούν αυτά που μας ε, εξηγήσατε και θα μείνουν ικανοποιημένοι. Όχι. Είστε επίτροπος αρμόδιος για τη δημόσια υγεία. Υποτίθεται ότι ε, προστατεύετε ε, τους καταναλωτές. Πώς έρχεστε και μας λέτε ότι δεν χρειάζεται και το γιατί είναι πανάκριβη και περίπλοκη. Τα δικαιώματα των πολιτών πού είναι. Ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην υγεία. Το θέμα δεν είναι η επισήμανση, ούτε θα μας γλιτώσει η ετικέτα. Εντάξει, καλή είναι η συμφωνία και σημαντική με τις Ηνωμένε Πολιτείε, λέω. Αλλά είναι πολύ περιοριστική η νομοθεσία μας για το τι μπορεί να παράγεται ε, στην Ευρώπη, ενώ αφήνουμε τις θύρες ορθάνικτες για παραγωγές τρίτων χωρών. Ο Chris Davis. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με το ηθικό και τη διδεντολογία και τα τρόφιμα. Αυτό που με ανησυχεί είναι η ευημερία των ζώων. Και είπατε 9 στα 10 κλωνοποιημένα ζώα δεν επιβίωσαν. Εκπροσωπώ ε, μια Βρετανική οργάνωση ε, για ε, την ευημερία των ζώων. Έχουν σε αυτά τα ζώα, προβλήματα στην αρτηριακή τους πίεση και ε, άλλα και είναι και πιο μικρό σώμα σε σχέση με τη μητέρα τους. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε λίγο αυτά τα θέματα της υγείας των ζώων και της ευημερίας και πώς θα ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε δεδομένων των ε, σημερινών καταστάσεων και εξελίξεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορτίνες Γκουτιέρες. Εγώ θα σας πάω σε άλλη κατεύθυνση. Όταν απορρίφθηκε η συμφωνία για την επισήμανση από το Συμβούλιο ε, τώρα εγώ δεν θέλω να σας κάνω κατά μέτωπο επίθεση, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά τότε υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις ετικέτες, διότι τεχνικά, όπως ήταν το σύστημα αναπαραγωγής, δεν μπορούσε να αποδείξει κανείς την κλωνοποίηση σε μία, δύο και τρεις γενιές πίσω. Και πάνω από 50 χρόνια ε, εισάγουμε σπέρμα από τις Ηνωμένε Πολιτείες που δεν ξέρουμε αν είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά κλωνοποίησης. Και από ό,τι φαίνεται επίσης τα κλωνοποιημένα ζώα από την πρώτη γενεά μοριακά δεν μπορούν να ανοιχνευθούν από την ε, μοριακή ανάλυση αν είναι κλωνοποιημένα ή όχι. Ενώ είναι. Το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο φαίνεται εδώ. Εμείς οι πολιτικοί έχουμε κάθε δικαίωμα ε, να λαμβάνουμε θέση με βάση την κοινή γνώμη ή την αίσθηση του κόσμου. Αλλά ρωτώ κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι έχει μεταφερθεί σε άλλο πεδίο το θέμα. Γίνεται ένα τεράστιο εμπόριο ε, ε σπέρματος από μια χώρα σε άλλη, εδώ και 50 χρόνια για τη σπερματέγχυση, ε, για τέτοιου είδους αναπαραγωγή και επιπλέον τεχνικά δεν είναι εύκολο να αποδείξει κανείς με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι λέει το έγγραφο και τι τεχνικοί λόγοι υπάρχουν, οι επιστημονικοί. Εγώ το ρωτάω αυτό για να έχετε αποφασίσει ως εξής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Επίτροπος παρακαλώ για να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων που ήταν επίσης πολύ άριθμες. Sorry, I have to come back on... Να επανέλθω σε κάποιες έννοιες. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις με διαφορετική έννοια. Αναφερθήκατε σε τρόφιμα από κλόνους. Τρόφιμα από κλόνους. Αυτό απαγορεύεται. Όχι, το λέω γιατί πρέπει να υποθεί. Συμφωνώ με την κυρία Ροτ Μπέρεντ ότι δεν είναι θέμα ασφάλειας τροφίμων. Υπάρχουν ε, κάποιες εμφιβολίες για το θέμα της ασφάλειας τροφίμων. Εδώ όμως δεν είναι θέμα ασφάλειας τροφίμων. Από πολιτικής απόψεως μπορεί να μου πείτε όμως ότι υπάρχει υπόνοια ότι είναι θέμα ασφάλειας των τροφίμων. Μπορεί να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να αγνοήσουμε την τεχνική γνώμη τη γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων και με το βλέμμα μας τραμμένο προς ε, τους πολίτες και με μια σχετική δημαγωγία να αναφερθούμε και στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και να πάρουμε μια άλλη απόφαση. Δεν είναι πάντα οι πιο δημοφιλείς αποφάσεις και οι πιο ορθές. Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα ασφάλειας των τροφίμων παρόλο που το κοινό μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το θέμα αυτό και κάποια άλλα επιχειρήματα βεβαίως. Ναι, όμως ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει, θέλει να γνωρίζει αν κάτι προέρχεται όχι άμεσα από κλωνοποιημένο ζώο, αλλά από κάποιο ζώο που προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο, δηλαδή από γόνους κλωνοποιημένων ζώων. Εξού και η πίεση για σήμανση. Αναφερόμαστε λοιπόν στην σήμανση και δεν αναφερόμαστε σε κλωνοποιημένα ζώα, αλλά σε ζώα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, από τους απογόνους. Και πού σταματάει κανείς, στην πρώτη γενιά, στην δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη γενιά. Όσον αφορά το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων, της ευμερίας των ζώων, ναι, εδώ το θέμα αυτό μας αφορά, ιδιαίτερα όσον αφορά την τεχνική κλωνοποίηση, καθότι πολλές φορές δημιουργούνται τερατογενέσεις σε κλωνοποιημένα ζώα, αλλά και όσον αφορά την ε, αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου. Δηλαδή πολλές φορές το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ χαμηλό, υπάρχει λοιπόν κακομεταχείριση ζώων, τα ζώα υποφέρουν και υπάρχει ε, και το θέμα της αποτελεσματικότητας. Μπορώ εδώ να σας πω ότι στην Επιτροπή δεν υπάρχει η πίεση ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα όποιες και να είναι οι συνέπειες. Όμως υπάρχει η πολιτική βούληση και η ιδέα ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, η TTIP, ε, πρέπει να συναυθεί. Ο αρμόδιος επίτροπος για τη διαπραγμάτευση αυτή σίγουρα έχει κατά νου ότι μία συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Τι διακυβεύεται λοιπόν σε σχέση με αυτό το θέμα στην TTIP. Εμείς συνεισφέρουμε στο δικό μας τομέα για τα θέματα που είναι δικής μας αρμοδιότητας, για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων. Επαναλαμβάνω ότι τα... οι Ηνωμένε πολιτείες πρέπει να δεχθούν τα παστηριωμένα προϊόντα μας και εγώ πάντα λέω ότι πίστευα ότι ο Παστέρ είναι Γάλλος, Ευρωπαίος. Γιατί λοιπόν το παστεριωμένο γάλα δεν είναι αρκετά παστεριωμένο για τους Αμερικανούς. Βεβαίως το θέμα του βόηου κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε ότι τόσα χρόνια μετά το θέμα της πογκόδους ε, εγκεφαλοπάθεια συνεχίζεται αυτή η απαγόρευση. Βέβαια πρέπει να περάσει και από το Αμερικανικό Κογκρέσο, όμως η απόφαση είναι πλέον σαφής. Θα έρθει η απαγόρευση για την εισαγωγή ευρωπαϊκού βοηουκρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των λαχανικών και των φρούτων και φυσικά σε καμία περίπτωση δηλαδή εδώ ότι εμείς θα υποχωρήσουμε σας αναφέρω απλώς ποια είναι τα ανοιχτά ακόμα θέματα. Υπάρχει βεβαίως και ο κανονισμός για τους, μη, ε, για τους γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Σαφώς και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν αντιμετωπίζουν το θέμα των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με τον ίδιο τρόπο. Και όταν αναφέρομαι στις δύο όχθες του Ατλαντικού υπάρχει βεβαίως και η Λατινική Αμερική. Έχουμε λίγο χρόνο, λέω. Ο Πρόεδρος για συμπληρωματικές ερωτήσεις αν υπάρχουν, να αξιοποιήσουμε το χρόνο. Ήταν όλοι οι συνάδελφοι σύντομοι. Α, τώρα αρχίζουν και σηκώνονται χέρια βλέπω. Η κυρία Παρβάνοβα, παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Μια βλακώδη ερώτηση θέλω να κάνω. Έχουμε μια απαγόρευση για την κλωνοποίηση των ζώων, αλλά παράλληλα θέλουμε να επισημαίνουμε τα τρόφιμα από απογόνους. Γιατί χρησιμοποιούμε τα κλωνοποιημένα ζώα και γιατί χρησιμοποιούμε τους απογόνους τους. Εάν απαγορεύουμε την κλωνοποίηση, γιατί επισημαίνουμε τους απογόνους. Νομίζω είναι παράλογο, δεν έχει νόημα. Θα έχει νόημα, έχει νόημα για την βιομηχανία, τον κλάδο. Αλλά μου φαίνεται ότι λέμε ψέματα στους πολίτες. Ε, απαγορεύουμε τους κλόνους, αλλά επιτρέπουμε τους απογόνους των κλόνων. Πώς μπορούμε να το πλασάρουμε αυτό στον κόσμο που σε τέσσερις μέρες θέλουμε να μας ψηφίσουν θα πρέπει να δοθεί μια λογική εξήγηση. Γιατί αυτή που προτείνεται δεν πρέπει να τους πείσει. Δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα Μακάβαν. Δεν με καταλάβατε. Εγώ δεν μίλησα για την ασφάλεια των τροφίμων. Μίλησα για τα θέματα ευημερία των ζώων. Γιατί έλεγα, ποιο ήταν το επιχείρημά μου. Αν πούμε κοιτάξτε, εμείς έχουμε δίκιο ηθικά. Ε, απαγορεύουμε τους, κλο, τους κλόνους γιατί είναι ε, ας πούμε κοινικό και σκληρό. Ε, τότε είναι λάθος να επιτρέπουμε την εισαγωγή σπέρματος από τις ΗΠΑ για να υποφελούμαστε στην παραγωγή τροφίμων από αυτό. Και η Κομισιόν μιλάει τώρα για τα έμβρια. Δεν μιλάει για αναπαραγωγικό υλικό. Υποτίθεται ότι κάνουμε κάτι για το πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι μοιάζει ε, η στάση μας. Ο κόσμος το καταλάβει. Είναι ε, σκληρό και δεν θα το κάνουμε τίποτα και δεν θα κάνουμε τίποτα στην Ευρώπη ή θα το δεχτούμε. Αλλά ας μην ε, προσποιούμαστε ότι έχουμε τόσο υψηλά πρότυπα ευημερία των ζώων, ε, απαγορεύουμε τους κλόνους αλλά επιτρέπουμε την πρακτική να συνεχίζεται από την πίσω πόρτα. Ευχαριστώ κύριε Ροτ Μπέρεντ. Γιατί θα πρέπει να υποκρίνεται κανείς εδώ, οποιοδήποτε, ότι μας ενδιαφέρει η ευημερία των ζώων. Δεκάρα δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολόκληρη. Ίσως εσείς λίγο κύριε Επίτροπε, αλλά είστε ο μόνος. Κανένας άλλος δεν ξέρω, καμιά φορά κανένας άλλος συνάδελφός σας, από καιρού καιρό, όχι συνέχεια. Ας είμαστε ειλικρινεί, βλέποντας τις δύο προτάσεις, εκεί που έχουμε ε, συναπόφαση είναι πάρα πολύ απλή, ε, ανόητη, απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά, ε, Μα χιλιάδες ε, ευρώ ε, κοστίζει να κλωνοποιήσεις ένα ζώο. Ποιος θα σκεφτεί να το σφάξει, να το κάνει τρόφιμο. Δεν συμφέρει αυτό. Μιλούμε για τους απογόνους και λέτε «Α, από τρίτες χώρες μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά» και τα και τα γιατί δεν γράφεται πραγματικά αυτό που εννοείται να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι δεν μας πειράζει να έχουμε προϊόντα αποκλωνοποιημένα ζώα, από γόνους, από τις Ηνωμένε Πολιτείε στην ευρωπαϊκή αγορά. Περί αυτού πρόκειται. Και θα πρέπει να βεβαιωθούμε απολύτως ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες τα γνωρίζουν. Και να δω μια κυβέρνηση που τολμάει να συμφωνήσει για το TTIP. Θα ε, την τορπιλήσουμε και ε, ε, είναι μόνο για αυτό το λόγο. <laughs> No, Mr. Stevenson. Ο κύριος Στίβενσον. I'm grateful to Linda. Είμαι ευγνώμων προς την ε, Λίντα και στην Ντάγμαρ γιατί ε, διευκρίνησαν τι ζητάει η Επιτροπή. Η συνέντευξη ποια είναι. Να απαγορεύσουμε όλα τα κρέατα, όλα τα γαλακτοκομικά και όλα στις αγωγές ε, σπέρματος από την Αμερική. Τελικά αυτά δεν λέτε. Γιατί στην Αμερική δεν έχουν κανέναν έλεγχο για την κλινοποίηση, δεν έχουν η θυλασιμότητα. Επομένως, τι μας λέτε, αν θέλουμε επισήμαση, δεν υπάρχει περίπτωση να συμμορφωθούν οι Αμερικάνοι. Βασικά βάζετε ένα φραγμό στο εμπόριο, θα ξεκινήσει ένα εμπορικό πόλεμο, Ντάγμαρ. Αν πας... Και πει, ας πούμε, οι Αμερικάνοι θα απαγορεύσουν τα δικά μας προϊόντα. Θυμάμαι θυμάμαι τον πόλεμο τη Μπανάνα. Ε, βάλαν οι Αμερικάνοι τότε, πήραν ένα κατάλογο από δικά μα προϊόντα και βάλανε χ σε διάφορα, με τυχαίο τρόπο. Αυτό ήταν ο εμπορικό πόλεμο μέχρι να τον επιλύσουμε. Τυχαία απαγόρευση ε, προϊόντων μα. Αυτό θα κάνει και η Αμερική, θα έχει πλήρη απαγόρευση. Γιατί οι Αμερικάνοι τόσοι άλλους επιτρέπουν την πλωνοποίηση, δεν έχουν ειχνασιμότητα και αυτό σημαίνει. Αν θέλει να προσπαθήσει να βρει από του απογόνου των κλωνοποιημένων ζώων, ούτω ώστε να βάλει την επισήμαση να κλωνοποιήσει, είναι αδύνατο να το κάνουν οι Αμερικάνοι, γιατί δεν μπορούν. Γιατί στην πραγματικότητα λοιπόν τι κάνετε έτσι με, αυτή την, ε, με τα επιχειρηματά σα, απαγορεύετε εισαγωγές από, από την Αμερική. Έχω την αντίδραση της Dagmar Roth Parent, γιατί αναφερθήκατε προσωπικά και μετά η, κυρία Κάντενμπαχ να τελειώσουμε για να απαντήσει ο Επίτροπος. Ε, εγώ νομίζω ότι ξέρω τι λέω. Όταν κάναμε για τα νέα τρόφιμα την πρώτη νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα, θελήσαμε επισήμαση και είπαν οι Αμερικανοί, δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε γιατί εμείς τα ανακατεύουμε όλα μαζί ε, σε πολύ μεγάλα βαγόνια και τα ε, μεταφέρουμε. Ε, ωραία, άμα δεν μπορείτε να τα διαχωρίσετε, τους είπα εγώ, να κολλήσετε παντού ετικέτες μεταλλαγμένα. Και ό, του θαύματος ξαφνικά μπορέσανε. Και ξέρω τι λες όταν μιλάς για εμπορικό πόλεμο. Θυμάμαι στις Ηνωμένε Πολιτείες χρησιμοποιούν ακόμα πέντε ορμόνες για το βόηο ε, κρέας, για τα βοηδή μάλλον, και οι περισσότεροι επιστήμονες λένε ότι τρεις από τις πέντε είναι καρκινογόνες και προκαλούν και ε, προβλήματα ε, σε αγόρια 14 με 16 ετών, θηλυκοποίηση και τα, ε, καταφέραμε να τα βγάλουμε, τα υπόλοιπα τα κρατήσαμε. Και πήγαμε και σε ένα πάνελ για ε, τα καλλιντικά και άλλα στον ΠΟΕ. Γιατί είναι λόγος να το δεχτούμε αυτό. Ούτε ηθικά στέκει, ούτε από πλευρά υγεία στέκει. Γιατί θα πρέπει εμεί να διαπαιδαγωγήσουμε το λαό μας. Οι Αμερικανοί να το κάνουν. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα να απαγορεύσουμε, να λέει η ετικέτα τι έχει μέσα, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάντενμπαχ. Νομίζω η τελευταία πρόταση της Τάκμαρ τα λέει όλα. Ότι θα βρούνε λύση για την ετικέτα. They will be able to label. Και αυτό το επιχείρημα ότι θα μας κάνουν εμπορικό πόλεμο είναι εκβιασμός. Δεν θέλουμε να εξαφανιστούν από την αγορά αυτά, αλλά να γνωρίζουν οι καταναλωτές, να έχουν μια δίκαιη ευκαιρία να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θέλουν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα ή όχι. Και γι' αυτό χρειάζεται σήμανση. Και η σήμανση ε, είναι εφικτή. Δεν μπαίνουμε τώρα σε τέτοια επιχειρήματα ε, με το μαχαίρι στο λαιμό. Θέλουμε την ελευθερία των ε, καταναλωτών να αποφασίζουν με τα λόγου γνώσεως και αυτό σημαίνει και είναι ως προϋπόθεση η ετικέτα. Ναι, εδώ τελειώσαμε από τα μέλη της Επιτροπής και τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Θα πάρει το λόγο ο Επίτροπος για να κλείσει. Thank you Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και για να το πω έτσι κάπως ε, διπλωματικά για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την καλή έννοια. Το σημειώνω και θα διαβιβάσω και τα μηνύματά σας. Κοιτάξτε. Θα μπορούσα να πω ότι δεν κάνουμε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς στο TTIP για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως επιχείρημα, τι το είπα εγώ. Έχουμε κόκκινη γραμμή και έχουν και εκείνοι κόκκινες γραμμές. Αυτό με τις ορμόνες που είπε η κυρία ε, Ροτ Πέρεντ. Συμφωνώ απολύτως. Πώς μπορούμε να βάλουμε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας σε κίνδυνο για να υπάρξει ακόμα μια συμφωνία που είναι ε, όντως ε, σημαντική, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγάλων εμπορικών ε, συνασπισμών ας πούμε, αλλά όχι πάση θυσία και με κάθε τίμημα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να μην δυσκολεύει ο ένας τον άλλον. Βεβαίως έχουμε υπόψη μας και τη συμφωνία TTIP, αλλά όχι με κάθε τίμημα και σε αυτό το θέμα η πρόταση να μην ε, συμπεριληφθεί επισήμαση δεν είχε ως βάση το TTIP. Ευχαριστώ την κυρία Ροτ Μπέρεντ για τα σχόλιά της σχετικά ε, με το ενδιαφέρον μου για την ευημερία των ζώων. Να, όντως με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, γιατί εν μέρη είναι και στο χαρτοφυλακείο μου. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν ε, ενδιαφέρον άλλοι επίτροποι Ιδιαίτερα γιατί κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα. Σήμερα το πρωί ε, μίλησα σε μία συνάντηση στο Σαρλεμάνιε, σε μια γεμάτη αίθουσα για την ευημερία των ζώων και ενδιαφέρθηκαν πολύ μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την ευημερία των ζώων και είναι θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο και στην προεκλογική εκστρατεία ακόμα περισσότερο και στους 14 μήνες που είμαι επίτροπος έχουμε προσφύγει στο δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ε, συγκεντρώσει τις έγκυες ε, σίες ε, νέου τάβλους που δεν έχουν εγκρίνει την οδηγία για τις Οτόκε όρνηθες και τα λοιπά ή που δεν έχουν εφαρμόσει τη γενικότερη νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης μπορούσε να αποφασίσει να παρατείνει την απαγόρευση ε, κυκλοφορία στο εμπόλιο καλλιντικών που έχουν χρησιμοποιηθεί οι πειραματόζωα ή να το αναβάλει. Εγώ στην ακρόαση μου είπα ότι δεν θα το αναβάλω ε, ε, να ε, επιβληθεί η απαγόρευση γιατί το έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και μετά από τόσο καιρό έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί αυτό που συμφώνησαν. Λοιπόν, Έχουμε θέματα ε, συζητήσει, έχουμε αρχίσει ήδη τις ε, προετοιμασίες για ένα γενικό νόμο πλαίσιο για την ευημερία των ζώων. Δυστυχώς θα είναι μετά τη λήξη της δικής μου και της δικής σας θητείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε λόγος για τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Επαναλαμβάνω, η τεχνική της κλωνοποίησης, τα τρόφιμα κλωνοποιημένα ζώα και η κυκλοφορία στο εμπόριο τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα δεν θα επιτραπεί αν εγκριθεί η παρούσα πρόταση. Πρόκειται για τρόφιμα από απογόνους κλωνοποιημένων που έχουν γεννηθεί και έχουν συλληφθεί προηγουμένως με τις κλασικές αναπαραγωγικές μεθόδους. Το ερώτημα είναι, θα πρέπει να επισημαίνεται τουλάχιστον η πρώτη γενεά για το νοπό βόηο κρέας από απογόνους πρώτης γενεάς κλωνοποιημένων ζώων. Το θέμα αυτό έχει αποφασιστεί τώρα. Και μπορώ να σας παραθέσω από τα πρακτικά της συνεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου ότι θα εκπονηθεί μελέτη σχετική που θα παραγγείλει η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας χωρίς να προεξοφλεί το αποτέλεσμα είτε της έκθεσης αυτής είτε της αποφάσεως της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν το λέω για παρηγοριά, απλώς για να σας πω ότι έχουμε αποφασίσει. Βεβαίως με την επιφύλαξη οποιοδήποτε ε, τροπολογιών που ενδεχομένως αργότερα ε, εισαγάγει το κοινοβούλιο στην πρόταση αυτή. Καλώς τελειώνει εδώ η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Είδατε από τις τόσες τοποθετήσεις ότι ε, πραγματικά μας καίει αυτό το θέμα. Ε, πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή μας που βλέπουν πολύ επικριτικά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφάνηκε ότι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών επίσης η πρόταση για την κλωνοποίηση είναι κάτι που μας πέφτει πάρα πολύ βαρύ σε πολλούς από εμά γιατί είναι μια πρόγευση για το τι θα γίνει και τι έπεται ενδεχομένως. Το είδατε και από τις επιμέρους συζητήσεις. Παρακαλώ αυτά τα πράγματα να πάρετε πάρα πολύ σοβαρά που σας είπαμε σήμερα. Να τα σημειώσετε, να τα διαβιβάσετε αρμοδίως και γνωρίζω ότι θα το κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, θα πρέπει να συμφωνήσει με τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Ακούσαμε σήμερα αριθμούς και στοιχεία πολλοί πολίτες έχουν τεράστιες επιφυλάξεις στην κλωνοποίηση και είμαστε και σε μια φάση που το Κοινοβούλιο στο τέλος της θητείας του ε, ε, ε, θα αναρωτηθεί για αυτά τα θέματα. Εγώ αν ήμουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός ε, ως προς την κλωνοποίηση. Και με μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον περιμένω τη συνέχεια και στο επόμενο κοινοβούλιο ε, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για το γεγονός ότι ήρθατε και παρουσιάσατε την πρόταση και την υπερασπιστή εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εύχομαι Καλό βράδυ σε όλους τους συναδέλφους και στον Επίτροπο. Προσεχή συνεδρία 17 Φεβρουαρίου. Το δικαίωμα στο νερό, η πρώτη πρωτοβουλία των πολιτών. Να έρθείτε όλοι, όσοι ήσασταν και σήμερα παρόντες, να έρθείτε και την άλλη Δευτέρα ε, και έχουμε την επίσημη συνεδρίασή μας 20 Φεβρουαρίου 9 με 12.30. Λήξη συνεδρίαση, καλό σας βράδυ.